για ε, ψήφισμα. Οπότε η ψηφορία θα γίνει μετά τη συζήτηση. Τελειώνει η συζήτηση για αυτό το θέμα και πάμε στο επόμενο ζήτημα. Πρόκειται για του ομαδικού τάφου των αγνωμένων τη Άσια στο χωριό Ορνήθη ή στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Προσοχή γιατί πιεζόμαστε τον χρόνο, έχουμε μείνει πίσω σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Επομένως, δεν θα επιτρέψω μπλε κάρτε για τη συγκεκριμένη συζήτηση. Και ούτε θα γίνει κάτσιδια για αυτό το θέμα, τόσο ώστε να μπορέσουμε να μείνουμε στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος για τις ψηφοφορίες. Ελπίζω ότι συμφωνείτε. Και τώρα, να δώσουμε το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Κέλλαμ. Επιμένω, θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός όσον αφορά την τήρηση του χρονικού πλαισίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ερώτημα των 2.000 και ενό αγνοούμενων Έλληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων είναι ανοιχτή πληγή για τις οικογένειες που θέλουν επιτέλους να μάθουν το τι έγινε αλλά και για την ειρνευτική διαδικασία στην Κύπρο και η Επιτροπή Αγνοουμένων εδώ πέρα κάνει πάρα πολύ σημαντικό έργο καθώς μέσω μαρτυριών βρίσκει μαζικούς τάφους και εξακριβώνει την ταυτότητα των νεκρών. Χρειάζεται λοιπόν ελεύθερη πρόσβαση και η Επιτροπή χρειάζεται επίσης την διακή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομική και πολιτική. Και στο πλαίσιο αυτό δεν αντιλαμβάνομαι γιατί μόλις εννέα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει την σύμβαση του ΟΗΕ για τους εξαφανισμένους θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι για αυτές τις βαρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μαριάς για ένα λεπτό. Πρόεδρε, το δράμα των οικογενειών των αγνοωμένων της Κύπρου μας έχει όλους κυριολεκτικά συγκλονίσει από τα νεανικά μας χρόνια. Χιλιάδες Ελληνοκύπριοι εδώ και 41 χρόνια αγνοούνται όταν τον Ιούλιο του 1974 τα τουρκικά στρατεύματα εισέβαλαν παράνομα στην Κύπρο και κατέλαβαν το 37% του νησιού όλοι αυτοί οι αγνοούμενοι δολοφονήθηκαν από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους σε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν στρατιωτικές για να εξαφανιστούν τα ίχνη τους. αλλά και όταν εντοπίζονται ομαδικοί τάφοι από τις προσπάθειες της επιτροπής αγνοωμένων όπως είναι και η περίπτωση του ομαδικού τάφου των αγνοωμένων της Άσιας που ανακαλύφθηκε στο χωριό ορνήθη και τότε τα τουρκικά στρατεύματα προσπαθούν ξανά να εξαφανίσουν τα ίχνη τα ψηφίσματα του οηε για τους κύπριους αγνοούμενους είναι δεκάδες. κόλαφος για την τουρκία είναι επίσης και οι καταδικαστικές αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ζητούμε λοιπόν να γίνει δεκτό το ψήφισμα για τους αγνοωμένους της κύπρου και της ασίας με το οποίο καλείται ο τουρκικός στρατός και η τουρκία να η για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην ελληνική τραγωδία και ο Σοφοκλής το 442 π.Χ. αναφέρθηκε στην Αντιγόνη στην ιστορία αυτή της αδερφής που ήθελε να κάνει τα πάντα προκειμένου να μπορέσει να θάψει τον αδερφό τη μετά το θάνατό του. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ίδια τραγωδία στην Κύπρο όπου μητέρε και πατεράδες όπου αδέρφια όπως και Αντιγόνη κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν τα λείψανα των αγαπημένων τους. Και δεν έχει λυθεί ακόμα από το 1974 η υπόθεση αυτή. Γι' αυτό τώρα οι αρχές πρέπει να κάνουν τα πάντα, στα κατεχόμενα, να βρεθούν τα λείψανα, να εντοπιστούν τα θύματα και να μπορέσουν να θάψουν τους αγαπημένους τους οι άνθρωποι εν ειρήνη. Ο κύριος Καρό, ένα λεπτό. Χώρα. Για 2.000 είναι γνώμενοι από τον πόνο 1974 και η συγγενείς δικαιούνται να μάθουν τι έγιναν οι αγαπημένοι τους. Τώρα όμως κινδυνεύουν μέχρι το θάνατό τους να μην έχουν μάθει τι έγινε. Θα πρέπει να πέσει φως αυτή την υπόθεση. Θα πρέπει ακριβώς να ασχοληθούμε με την υπόθεση και να ξεκινήσει μια διαδικασία συμφιλίωσης στην Κύπρο. Υπάρχει μια επιτροπή που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά αλλά χρειάζεται συνεργασία και με τις αρχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι κάνει η Τουρκία. Ε, την οποία χρηματοδοτούμε υπάρχουν και οι διαδικασίες προενταξιακές. Άρα θα πρέπει να πιέσουμε την Τουρκία ούτως ώστε να βοηθήσει και να κάνει κάτι για αυτή την υπόθεση. Κύριε Χατζηγεωργίου, 1,5 λεπτό. Συνάδελφοι, εδώ και μερικά χρόνια δεκάδες ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι επιστήμονες αλλά και απλοί πολίτες εργάζονται στην προσπάθεια να βρουν τα οστά των νεκρών της κυπριακής τραγωδίας και αυτό νομίζω ότι αποτελεί μια πράξη που αναδεικνύει ε, την ανθρώπινη φυλή. Το να εργάζεσαι δηλαδή στο να βρεις τους τύπους της ιστορίας και να ανοιχνεύσεις τα βήματα της και τον πόνο των ανθρώπων και των συγγενών τους ούτως εχόντων των πραγμάτων την ίδια ώρα είναι πράξη ντροπή η μετακίνηση και η εξαφάνιση οστών από μαζικούς τάφους. Μια πράξη ισοδύναμη σκέφτομαι κάποτε με την ίδια την πράξη της δολοφονίας. Θεωρώ λοιπόν σωστό να καλέσουμε την Τουρκία να πάψει αυτή την τροπιαστική ενέργεια, να δείξει τους τόπους της ταφής ε, των αγνοουμένων, των δολοφονηθέντων και να ανοίξει τα αρχεία της για να γνωρίσει η διερευνητική επιτροπή πού πρέπει να ψάξει. τέλος καλούμε το συμβούλιο να αυξήσει οικονομικά την ενίσχυσή του προς την διερευνητική επιτροπή προκειμένου αυτό το έργο να το διεξέλθεται κανείς όσο δυνατόν πιο εύκολα. ο αγώνας είναι αγώνας για την ανέβρεση των οστών όλων των νεκρών της κυπριακής τραγωδίας ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων γι' αυτό είναι που εξέφρασα την τιμή και την εκτίμησή μου προς τους ανθρώπους ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους που εργάζονται σε αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, Είναι απαραβίαστο ανθρώπινο δικαίωμα να σεβόμαστε τουλάχιστον το σώμα των νεκρών είναι η κληρονομιά της Αντιγόνης. Και βεβαίως όλοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πού έχουν ταφεί οι οικοί τους και να έχουν πρόσβαση στον τάφο τους. Και να ξέρουν πώς πέθαναν. Αυτό είναι το νόημα του ψηφίσματος αυτού. Υπάρχει βεβαίως εδώ πέρα η παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων και αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό είναι αναγκαίο αυτό το ψήφισμα. Μόνο έτσι θα υπάρξει η μνήμη και χωρίς τη μνήμη δεν υπάρχει μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να ισχύσει αυτό το οποίο αναφέρεται στην Αντιγόνη, ότι δεν έχουμε γεννηθεί για να μισούμε, αλλά για να αγαπάμε. Η κυρία Ιδεχοχάρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ένα έγκλημα πολέμου που διεκπράχθη το 1974 από τον τουρκικό στρατό εισβολή στην Κύπρο με μαζικές εκτελέσεις αδειλώτων, εχμαλώτων και αμάχων οι οποίοι ετάφησαν σε άγνωστου για χρόνια μαζικού τάφους τα κατεχόμενα εδάφη έρχεται ξανά στην επιφάνεια με αφορμή την τραγική περίπτωση των μαζικών τάφων που ανεβρέθησαν στο χωριό ορνήθη αλλά και σε άλλε περιοχέ. Στι περιπτώσει αυτέ, ο τουρκικό στρατό μετακίνησε τα οστά αμάχων δολοφονηθέντων από το χωριό Άσια σε άγνωστο μέρο, και δεν ανεβρέθησαν παρά μόνο ελάχιστα υπολείμματα οι μετακίνησει των οστών γίνονται για να μην εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου των θυμάτων. γι' αυτό ζητάμε από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να καλέσει την τουρκία να σταματήσει να συμπεριφέρεται ασεβώς προς τους νεκρούς να σταματήσει την ύβρη προς την ανθρωπότητα να σταματήσει τις μετακινήσεις των νεκρών από τους μαζικούς τάφους και να ανοίξει τα στρατιωτικά της αρχεία και τις λεγόμενες στρατιωτικές ζώνες προς διερεύνηση και απόδοση των νεκρών στις οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εδώ και 40 χρόνια η Τουρκία παραβιάζοντας κάθε αρχή ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου κατέχει μέρος της πατρίδας μας με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραγικές συνέπειες τόσο για τον λαό μας όσο για την Κύπρο αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο τραγική όμως πτυχή αυτού του κυπριακού δράματος είναι η πτυχή των αγνωμένων. Το ότι εδώ και 40 χρόνια υπάρχουν Κύπροι αγνοούμενοι είναι γιατί η Τουρκία και αυτό το κατεξοχή ανθρωπιστικό θέμα επιδεικνύει ένα απάνθρωπο και σκληρό πρόσωπο αρνείται να ανοίξει τα αρχεία του τουρκικού στρατού για να διερευνηθεί η τύχη του. Εκεί και όπου εντοπίζονται μαζικοί τάφοι αγνοωμένων, του χαρακτηρίζει κλειστή στρατιωτική περιοχή. Και το σημαντικότερο και το κυριότερο και το πιο αισχρό είναι ότι μετακινεί οστά αγνοωμένων όπω έγινε στην Άσσα για να εξαφανίσει τα ίχνη. Δυστυχώ αυτή είναι η Τουρκία. Αυτή είναι η Τουρκία που δεν σέβεται του νεκρού. Αυτή είναι η Τουρκία η οποία ουσιαστικά θέλει να γίνει χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η Τουρκία η οποία λαμβάνει προενταξιακή βοήθεια. Ε, Εμεί καλούμε να ληφθούν κυρώσει εναντίον τη Τουρκία για αυτό το ζήτημα. Παπαδάκη για ένα λεπτό. Ε. Κύριε Πρόεδρε, το ανθρώπινο δράμα δεν ξεχωρίζει φυλές και εθνοτικές καταγωγέ αυτό που γίνεται τώρα στο κατεχόμενο τμήμα της κύπρου είναι ένα δεύτερο έγκλημα απέναντι σε ολόκληρη την ανθρωπότητα αφού σαράντα χρόνια μετά το κατοχικό καθεστώς της τουρκίας μετακινείται οστά των αγνοωμένων προσπαθώντας να εξαφανίσει στοιχεία που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό τους. Σκεφτείτε τους συγγενείς των αγνοωμένων να αναρωτιούνται τι απέγιναν οι δικοί τους άνθρωποι σκεφτείτε να θάβουν ένα κομμάτι από το δάχτυλο ή ένα κομμάτι από το πόδι τους. Η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και οφείλουμε να καλέσουμε άμεσα την Τουρκία να συνεργαστεί για την πλήρη διερεύνηση της τύχης των αγνοωμένων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Εδώ δεν χωρούν πολιτικά παιχνίδια η τιμή των νεκρών είναι ό,τι πιο ιερό στην ευρώπη. δεν μπορεί να υποκρίνεται η ευρώπη για να εξυπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες. ένα λεπτό. Πρόεδρε, το 2011 ήμουν και εγώ συντάκτης μιας επιτυχούς δήλωσης για το έργο της Επιτροπής που ασχολείται με τους αγνοούμενους στην Κύπρο. Σήμερα το ψήφισμά μας θέλει μια παραπάνω έκκληση να κάνει όσον αφορά τους ομαδικούς τάφους στην Άσια όπου φαίνεται 106 αγνοούμενοι βρίσκονται μετά από δολοφονία το 1974. Τα λείψανά τους όμως έχουν μεταφερθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Η Τουρκία πολλές φορές έχει κριθεί και από το Διεθνές Δικαστήριο όσον αφορά τα εγκλήματά της στη Βόρεια Κύπρο. Είναι υποχρεωμένη να βοηθήσει να εντοπιστούν όλα τα λείψανα που παραμένουν ώστε να καταλάβουμε ποια ακριβώ ήταν η αιτία του θανάτου του. Μετά από 40 χρόνια δεν είναι δυνατόν να μην έχει κλείσει ακόμα αυτή η ιστορία και να μην μπορούν οι άνθρωποι να θάψουν του αγαπημένου του. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν όλοι οι ομαδικοί τάφοι, διακόπτει ο πρόεδρο, η κυρία Άντερσον για ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στην Κύπρο και την Ιρλανδία, γιατί εκεί δύο είναι νησιά, είναι διαιρεμένες χώρες, έχουν ξένη κατοχή και διένεξη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο να υπάρξει συμφιλίωση και αλήθεια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι η υπόθεση των αγνοουμένων είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν οι τουρκικές αρχές, οι οποίες δυστυχώς δεν διεξήγαγαν αποτελεσματική διερεύνηση και παραβιάζουν το άρθρο 2 της σχετικής σύμβασης. Επίσης ζητούμε να Πρέπει να λάβουμε επίση υπόψη μα τα κοινά σημεία που υπάρχουν ανάμεσα στη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να παραβιάζει το άρθρο 2 για δολοφονίε από το κράτο στη Βόρεια Ελλάδα. Ζητούμε λοιπόν συμφιλίωση στην Κύπρο και για να επιτευχθεί αυτό η Τουρκία πρέπει να αποκαλύψει την αλήθεια όσον αφορά του αγνοούμενου και σε σχέση με το έγκλημα τη μεταφορά λιψάνων που, με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν τουρκικέ αρχέ. Ο κύριο Καλστάλδο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Πάρα πολλά μπορεί να είναι τα πτώματα σε έναν κοινό ε, τάφο, αλλά πόσο βαθύ θα πρέπει να είναι ο τάφος ώστε να ταφεί εκεί πέρα η ιστορία και οι ευθύνε από αυτόν τον ε, τρομερό πόλεμο, από αυτή την τρομερή ιστορία που θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ε, βαθύ ο τάφος για να χωρέσει αυτό το πήγαινε και στην Άσα. Και βλέπουμε τώρα ότι είναι απελπισμένες οι οικογένειε για αυτό το οποίο έγινε για κάτι το οποίο θα πρέπει να λεληθεί έστω και αργά, ούτω ώστε να μπορέσουν να, να βρουν τους, το πτώμα των αγαπημένων του οι οικογένειε αυτές. Ε, είδατε πόσε καταδίκε έχουν γίνει, υποθεμένως επομένω όλε οι πολιτικέ πτέρυγες του Κοινοβουλίου να πιέσουν ούτω ώστε να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Πρόκειται για υποψήφια χώρα προ ένταξη, άρα θα έπρεπε να υπάρχει υπόσχεση, δέσμευση, συνεργασία και όχι αυτή η επονίδιστη σιγή. Το να μην κάνουμε τίποτα θα ήταν μεγάλο λάθος. Φεράν, ένα λεπτό. Ένα λεπτό κύριε Φεράν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή η τραγική περίπτωση του κοινού τάφου είναι το πρόσωπο το μακάβριο της ε, κατοχής της Κύπνου μετά 41 χρόνια. Είναι ένοχο το τουρκικό κράτος, αλλά είναι συνένοχοι και εκείνοι που κάνουν τις διαπραγματεύσεις της ένταξης εδώ και μια δεκαετία. Ο πρόεδρος του, ο πρόεδρος του Βελγίου, ο Φερχόφστατ και όλοι αυτοί οι οποίοι μαζί με τον Ερντογάν απεργάζονται την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο μία είναι η λύση σήμερα το να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις αυτές για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα λεπτό, Πόλτσακ. Ευχαριστώ και με τη σειρά μου να σας τονίσω ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Τουρκία έχει παραβιάσει δικαιώματα τα δικαιώματα εκείνων που έχασαν τους αγαπημένους τους. Η Τουρκία δεν απεζημίωσε ως όφιλε σύμφωνα με όσα έκρινε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται περί σκανδάλου. Η χώρα, η Τουρκία, έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όμως δεν αναγνωρίζει την Κύπρο. Αρνείται να καταβάλει τις δέουσες αποζημιώσεις στα θύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δίνει πολλά στην Τουρκία. Ε, Υπάρχουν τα χρήματα να κατεβούν θέση αποζημίωση. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Λόγω των εσωτερικών λόγω των συγκρούσεων και της τουρκικής κατοχής Έχουμε χιλιάδες ε, αγνώμενους. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα. Το 1974 πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι στην ε, περιοχή εκείνη. Έχουν υπάρξει πολλές ε, καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ακόμα αναζητούμε πληροφορίες. Πρέπει λοιπόν να απευθύνουμε μία έκκληση στους Τούρκους να κάνουν κάτι πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτή την ε, τραγική κατάσταση. εξαφανισμένη. εξαφανισμένοι ακόμα δεν έχουν ε, ταυτοποιηθεί και δεν έχουν άρα αναπαυθεί. Ζητάμε λοιπόν ε, και από τις δύο πλευρές να κάνουν κάτι. Ένα λεπτό κύριος Χρυσόγονος. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η συνεχιζόμενη έκτοτε κατοχή του 40% του νησιού συνιστούν καθεαυτές μείζωνος σημασίας παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τις οποίες η τουρκία έχει καταδικαστεί κατ' επανάληψη από το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου. αυτή η μείζον παραβίαση συνοδεύθηκε από ιδεχθή εγκλήματα πολέμου όπως η μαζική εκτέλεση 1.600 περίπου ελλήνων και ελληνοκυπρίων εχμαλώτων που λογίζονται ως αγνοούμενοι επί 40 χρόνια. Τα εγκλήματα εκείνα όχι μόνο δεν έχουν αναγνωριστεί και τιμωρηθεί, αλλά η τουρκική πλευρά επιδίδεται σε διαρκή προσπάθεια συγκάλυψής τους. Ένα επιμέρους επεισόδιο είναι η πρόσφατη μεταφορά οστών από την περιοχή της Άσκιας σε άλλη άγνωστη περιοχή στα κατεχόμενα. Είναι ντροπή για τον ευρωπαϊκό πολιτικό και νομικό πολιτισμό ότι γίνονται ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές από ένα... Carver James. Ευχαριστώ. Carver James για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσωπική τραγωδία από το να μην ξέρει κανείς τι απέγιναν οι οικοί του. Η Επιτροπή Αγνοωμένων που συστάθηκε πριν από 34 χρόνια μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιήσει 568 θύματα και από τις δύο κοινότητες για να μπορέσει ακριβώ να κλείσει κάποιες περιπτώσεις των 1443 Κυπρίων. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω πως έχει φτάσει η στιγμή για μια νέα προσέγγιση στο τραγικό αυτό ζήτημα. Θεωρώ πως η Κύπρος πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Νοτιού Αφρικής μετά το καθεστώς του Απαρχάιντ με το να φτιάξει μια επιτροπή αλήθειας και συμφιλίωσης για να διακριβωθεί η μοίρα και η τάφη των αγνοωμένων. Ίσως όχι μέσω των ε, γνωστών ε, διπλωματικών ομάδων. Κύριος Φουντούλης για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά για κάποιους ίσως είναι ελληνικά γράμματα τυπωμένα απλά σε χαρτί. στην πραγματικότητα όμως αυτά τα ονόματα αντιστοιχούν σε άνδρες που ήταν πατέρες παππούδες γη και εγγονοί. οι περισσότεροι κατάγονται από την άσια. η άσια και οι κάτοικοί τη βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα και της βαρβαρότητας των τουρκικών στρατευμάτων. αθώοι πολίτε εκτελούνται εψυχρό τι πρώτε ώρε μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής αιχμαλώτων τους επόμενους μήνες 84 άνθρωποι δεν γύρισαν ποτέ όλα τα εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπράξει τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και οι τουρκοκύπροι συνεργάτες τους και ιδίως αυτό που διαπράχθηκε στην κατεχόμενη Άσια παραμένουν ατιμόρυτα μέχρι σήμερα. Οι Τούρκοι για να καλύψουν τα εγκλήματά τους δεν σεβάστηκαν ούτε τους νεκρούς ασιώτες. Μετακίνησαν τα οστά από τους ομαδικούς τάφους και τα έριξαν σε πηγάδια και σκουπιδότοπους για να μην βρεθούν ποτέ. Όπως είναι ήδη γνωστό οι εκταφές το 2009 που έγιναν από τη Δέα επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες τα προβλήματα που προκύπτουν σε... Îl Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε να σας δώσω το λόγο πριν όμω από αυτό να κάνω μια έκκληση στου ε, συναδέλφους κάντε λίγη ισχύα για να ακούσουμε τον Επίτροπο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είπα ότι εκπρόσωπος και αντιπρόεδρο ε, Φεντερίκα Μογκερίνη μου ζήτησε να διαβάσω το εξής μήνυμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει την ανθρώπινη διάσταση των συνεπειών των τραγικών γεγονότων του 1963-64 και 1974 για τον πληθυσμό ολόκληρης της Κύπρου. Αναπάντητα ερωτήματα, ειδικά αυτά που αφορούν τους αγνώμενους, δεν επιτρέπουν σε πολλούς ε, Κύπρους ε, και από τις δύο κοινότητες ε, να αφήσουν πίσω το παρελθόν για τις οικογένειές τους λοιπόν έχει κρίσιμη σημασία το να ξέρουν ποια είναι η μοίρα των δικών τους. Γι' αυτό η Κομισιόν σκοπεύει να στηρίξει το έργο του ΟΗΕ και της ε, Επιτροπής Αγνοουμένων. Η Επιτροπή Αγνοουμένων έχει μια ανθρωπιστική εντολή και συνεισφέρει στην ε, ανακούφιση των αγνοουμένων των οικογενειών των αγνοουμένων και έχει αποδειχθεί ένα επιτυχημένο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και άρα συνεισφέρει στην συμφιλίωση, στην ίσο η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης της Επιτροπής Είναι μια συνολική συνεισφορά από το 2006 14,7 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία διαχειρίζεται η συνάδελφος κυρία Κρέτσου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο της Επιτροπής Αγνοωμένων και θα δώσει άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το 2015. Επίσης θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο για προηγούμενα χρόνια έδωσε επιπλέον χρηματοδότηση για την Επιτροπή των Αγνοωμένων και θα ήθελα εδώ πέρα να αποτίσω φόρο τιμής στους κυρίους ε, Παναγιώτη Δημητρίου, Ιωάννη Κασουλίδη Κλάμπτ και Μπουσουτήλ καθώς και στους νυν βουλευτές Μπέγκε, Θεοχάρους και Χατζηγεωργίου. Η Επιτροπή συμφωνεί πως περισσότερα πρέπει και μπορούν να γίνουν από όλους ε, τους ενδιαφερόμενους για να ξεκαθαρίσει η μοίρα όλων των αγνοωμένων. Ταυτόχρονα η κατάσταση περιπλέκεται καθώς ε, νέες πηγές πληροφοριών ε, πλέον λιγοστεύουν και δεν είναι προσβάσιμη η μαζική τάφη. Γι' αυτό θα πρέπει η Επιτροπή Αγνοωμένων να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά αρχεία και βεβαίως στις στρατιωτικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τακτικά ζητάει από την Τουρκία να συμμορφωθεί. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, η αγνώμενη είναι ένα ζήτημα ανθρωπιστικό. Αυτό, όπως και πολλά άλλα ζητήματα, δείχνει την ανάγκη για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει την επανάληψη των συνομιλιών υπό την αιγύδα του ΟΗΕ. Ξεκαθαρίσαμε την ετοιμότητά μας να βοηθήσουμε. Στηρίζουμε τις προσπάθειες του απεσταλμένου του ΟΗΕ, κυρίου Άιτε, και πρέπει να βρεθεί μια απάντηση και να στηρίξουμε και τις δύο κοινότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έχουμε 7 προτάσεις ψηφίσματος, η συζήτηση τελείωσε και ακολουθούν οι ψηφοφορίες. Înainte de a trece la votare, am o solicitare din partea... Αλλά από την ΚΟΕ, η κυρία Φορέντζα έχει κάτι να ρωτήσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χθες, όπως και αναφέρθηκε στην Ολομέλεια, είχαμε τον θάνατο 300 ανθρώπων στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα. Είναι η πολλωστή τραγωδία